Um, right, good morning. Well, I have the rapporteur and the S&D and ALDI shadows for the for the first uh, matter. Uh, I have. Καλημέρα σας. Δεν γνωρίζω αν οι υπόλοιποι σκιώδεις εισηγητές θα, εισηγητές θα έρθουν. Ωστόσο, ε, μία εισηγήτρια σκιώδης πρέπει να προεδρεύσει στη δική της επιτροπή Γι' αυτό και προτείνω να αρχίσουμε ευθύ αμέσω. Είναι λίγο μετά τι 9 και είμαι σίγουρη ότι και ο εισηγητή και οι σκιώδει εισηγητέ γνωρίζουν το ιστορικό υπόβαθρο τη ε, πρότασης αυτής. Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση τον Ιούνιο του 2012. Από πλευράς διαδικαστικής περιπλέκεται το πράγμα, διότι χρειαζόμαστε απόλυτη συμβατότητα με την έκθεση Γκοζέση για το διπλό νομοθετικό πακέτο. Η Επιτροπή όμως δεν προτείνει την ενημέρωση εκείνης της πρότασης και βασική ιδέα είναι ότι θα σημειωθούν ορισμένες αλλαγές με τη, με τη διαδικασία στο Συμβούλιο. Η Επιτροπή ενδιαφέρεται για όσα έχουμε εμείς να πούμε είναι μια διαδικασία στην οποία μπορούμε να απαντήσουμε καταφατικά ή αποφατικά, ναι ή όχι, μόνο. Αλλά μπορούμε ήδη να ανοίξουμε κάποια από τα χαρτιά μας για το προς ποια κατεύθυνση θέλουμε να πάρουμε και ελπίζουμε να τα λάβουν υπόψη τους αυτά η Επιτροπή και το Συμβούλιο. Αυτά λοιπόν από πλευράς διαδικασίας να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια κυρία Χιούμπνερ. Ευχαριστώ Σάρων. Θα θυμάστε πράγματι το ιστορικό υπόβαθρο, θα θυμάστε ότι από το 2002 είχαμε νομοθετήσει ένα τέτοιο μέσο παροχής οικονομικής βοήθειας στα κράτη-μέλη που δεν είναι μέλη της ε, ζώνης του ευρώ, αλλά το, τα οποία κράτη-μέλη ενδεχομένως θα είχαν δυσκολίες στην εξωτερική τους χρηματοδότηση. Αναφερόμασταν κυρίως στη Λετωνία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία. Το 2002 μάλλον εννοεί η ομιλήτρια και όχι το 1992. Από εκεί και πέρα είχαμε κρίση στη ζώνη του ευρώ, όπως γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια. και δεν είχε προβλεφθεί τίποτα για τις χώρες που δεν ήταν ε, ε, μέλη της ζώνης του ευρώ. Επιτέλους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει κάποιες προσαρμογές στον υφιστάμενο κανονισμό. Επιτέλους έχουν προβλεφθεί προτάσεις για να μπορούν αυτά τα κράτη-μέλη να έχουν οικονομική βοήθεια και ο κανονισμός αυτός ενημερώνεται λοιπόν υπό το πρίσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης και προβλέπονται και νέα εργαλεία από πλευράς γραμμών πίστοσης ή από πλευράς δανείων. Επί της διαδικασίας, εν συντομία να πω ότι δύο είναι οι βασικές μας δυνατότητες. Μία έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας καταρχάς. Εμείς ως Επιτροπή Οικονομικών υποθέσεων και βεβαίως όλο το Κοινοβούλιο μπορεί να συμβάλλει στη σύνταξη αυτής της έκθεσης ίδιας πρωτοβουλίας για το ποιες προσδοκίες έχουμε έναντι Συμβουλίου και κρατών μελών ως προς τις προτάσεις της Επιτροπής ή αν δεν υπάρχει περιθώριο για την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας, περιμένουμε να μας απαντήσουν, μπορούμε να καταλήξουμε σε ψήφισμα της Επιτροπής μας ή και σε επιστολή ενδεχομένως. Ας ελπίσουμε όμως ότι το δίλημα θα ταθεί μόνο μεταξύ έκθεσης ίδιας πρωτοβουλίας και ψηφίσματος. Από πλευράς χρονικής συγκυρίας τώρα, ελπίζω το αργότερο μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου να έχουμε ένα πρώτο σχέδιο της έκθεσης, το οποίο να εξετάσει η Επιτροπή μας των Οικονομικών Υποθέσεων στα τέλη Ιανουαρίου και άρα να ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Απριλίου. Η πρόκληση που υψώνεται μπροστά μας είναι να δούμε τα στοιχεία της έκθεσης του κυρίου Γκοζές, τα οποία θα πρέπει να προσθεθούν σε αυτόν εδώ το κανονισμό. Προτείνω στην Επιτροπή μας να εξετάσει και κάποια επιπρόσθετα ζητήματα, να δούμε κατά πόσο μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε. Έχουμε ήδη συναντηθεί με τους συναδέλφους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρακολουθούν ε, την έκθεση Γκοζές και τις αλλαγές που υπησέρχονται εκεί και ανέφεραν ότι βεβαίως θα πρέπει να αναθεωρηθεί ο κανονισμός υπό το φως των καινοτομιών που εισήγαγε το Κοινοβούλιο διαμέσου της έκθεσης Γκοζές και ελπίζουμε ότι θα ε, λάβουν υπόψη τους και νέα ζητήματα που θα έχουν ε, προκύψει μετά από τη δουλειά που έχω κάνει εγώ με τους εισηγητές. Τώρα, προκειμένου να έχουμε ένα παιχνίδι επί ίσης όρης μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ και των χωρών που είναι εκτός ευρώ, μας ενδιαφέρουν τα προγράμματα μακροοικονομικής προσαρμογής, γιατί ε, αυτά θα αντικαταστήσουν διάφορα διάφορα βήματα και στάδια παρακολούθησης και εποπτείας. Και αυτό είναι σημαντικό. Ε, αναφερόμαστε στην ενισχυμένη εποπτεία για τα κράτη-μέλη που θα λάβουν βοήθεια για λόγους πρόληψης και αναφερόμαστε και στη διαφάνεια και στη λογοδοσία ως προς το ρόλο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων σε όλη αυτή τη διαδικασία και ως προς τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάζει ε, όλα τα στοιχεία της διαδικασίας και θα μας ενημερώνει. Περιμένουμε διαφάνεια παντού και αναφερόμαστε και σε κάποια ίσονο σημασία ζητήματα σε σχέση με το σύνολο της διαδικασίας, αλλά έχουν συμπεριληφθεί χάρη στην έκθεση του κυρίου Γκοζέσου. Υπάρχουν κάποια θέματα ωστόσο για τα οποία θα ήθελα να τοποθετηθώ. Στην έκθεσή μας αναφερόμαστε στην ασάφεια ορισμένων ορισμών και ορισμένων στοιχείων. Π.χ. η μεταβατική διαδικασία από το ένα μέσο ενίσχυσης και βοήθεια στο άλλο ή κάτι που πρέπει να μας προβληματίζει περισσότερο είναι η ανάγκη των κρατών μελών που είναι εκτός του ευρώ να ζητήσουν άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν απευθύνονται στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κάτι το οποίο δεν ισχύει για την Ευρώπη. Και επίσης υπάρχουν και κάποια θέματα για την αναλογικότητα, την επικουρικότητα και το καθεξής. Κάτι που δεν μπορούμε να αλλάξουμε, το ξέρω αυτό, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να αρχίσουμε να το θέτουμε, είναι να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία ώστε και για τις χώρες που δεν είναι μέλη του ευρώ να υπάρχει αυτό το οποίο ονομάζουμε fiscal backstop. Δηλαδή ένα σύστημα, εν πάση περιπτώσει, επιθεώρησης. Δηλαδή, ε, αυτό θα σήμαινε ότι οι χώρες εκτός ευρώ ε, αν δεν συμμετέχουν τουλάχιστον θα ε, μπορούσαν να παρίστανται στον ενίο εποπτικό μηχανισμό. Σε αντίθεση με τις χώρες που έχουν το ευρώ δεν θα έχουν αυτό το fiscal backstop. Και θα πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Να υπάρχει κάτι ανάλογο. Και ελπίζω αυτό να ε, τύχει υποστήριξη στο συντομότερο δυνατό. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν όρια ως προς την οικονομική βοήθεια, διότι αυτή η οικονομική βοήθεια η οποία έχει ως εχέγγυο τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό έχει ένα όριο 50 ή 60 δις ευρώ, ενώ για παράδειγμα για την ανακεφαλοποίηση των ε, τραπεζών π.χ. Ε, θα χρειαζόντουσαν πολύ περισσότερα κονδύλια. Υπάρχουν δηλαδή κάποια θέματα και από τη στιγμή που θα πρέπει να υιοθετηθεί η συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ώστε να μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό το μηχανισμό και οι χώρες που δεν έχουν το ευρώ και να μπορούν να συμμετάσχουν στο σκέλος του μηχανισμού που αφορά στην ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, τότε θα πρέπει να εξετάσουμε άλλες επιλογές. Π.χ. να δημιουργήσουμε ένα νέο ταμείο διαμέσου της διακυβερνητικής συνθήκης ή κάποια άλλα τα οποία ε, θα συμπεριλάβω στην έκθεσή μου. Είχαμε λοιπόν μια πρώτη συνάντηση μεταξύ εμού και των σκιωδών συζητητών και ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε να έχουμε ένα σχέδιο έκθεσης μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου ώστε να κινηθεί η διαδικασία αρκετά γρήγορα ή τουλάχιστον παράλληλα με τη διαδικασία της έκθεσης Γκοζές. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Έρχομαι στους σκιώδεις συζητητές τώρα. Ο Σάβιν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι και εμείς βεβαίως πάντοτε μπορούμε να σχολιάσουμε ε, ε, αυτή, αυτό το φάκελο, παρόλο που γενικά έχουμε συνένεση και υπάρχει συνένεση, ε, συμφωνώ με την πρόταση για την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας ή τουλάχιστον ψήφισμα. Μετά την προκαταρκτική συζήτηση που είχαμε την εισηγήτρια μπορώ πράγματι να επιβεβαιώσω ότι κινούμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Με την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση είναι αληθές ότι τα μέρη τα κράτη-μέλη που δεν είναι στο ευρώ δεν είχαν μέχρι τώρα ε, χρηματοδοτικά εργαλεία στη διάθεσή τους αρκετά και τώρα θα έχουν περισσότερα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μπορεί να δίδεται οικονομική βοήθεια ε, και να συμπεριληφθούν αυτά τα κράτη, να τους δίδεται οικονομική ε, βοήθεια στα κράτη που δεν είναι στο ευρώ. από εκεί και πέρα το σύνολο των 50 δις ευρώ δεν αλλάζει και εγώ νομίζω ότι είναι καλό αυτό. Θέλω όμως να θέσω το εξή θέμα. Από τη στιγμή που θέλουμε να ευθυγραμμίσουμε τις συνθήκες και τις διαδικασίες για την παροχή οικονομικής βοήθειας που ισχύουν για τα κράτη του ευρώ στα κράτη που δεν είναι στο ευρώ, τότε τουλάχιστον να μπορούν να αξιοποιήσουν και οι δύο ομάδες κρατών τις ίδιες γραμμές πίστοσης. Ξέρω ότι αυτό είναι αδύνατο γιατί είναι πολιτικό το ζήτημα. Ωστόσο θέλω να το θέτω αυτό το ζήτημα, να διερευνηθεί κατά πόσο μπορεί να βρεθεί μια νομικώς εφικτή λύση. Περιμένω τώρα ε, να δω το χρονοδιάγραμμα, διότι ε, αυτό... Ε, διότι έχουμε κάποιους περιορισμούς. Δεν ξέρουμε ακόμα αν τελικά θα έχουμε έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας ή ψήφισμα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι το κείμενο θα είναι πολύ καλό. Ευχαριστώ εκ μέρους του Άλντε ο κύριος Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Ντανούτα Χιούμπνερ. Είχαμε μια πρώτη συζήτηση και εγώ τουλάχιστον έμαθα αρκετά. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό το γεγονός ότι αναθεωρείται αυτός ο κανονισμός και συμμερίζομαι τις απόψεις που εξέφρασε η κυρία Τανούτα Χιούμπνερ. Θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε τις απόψεις μας, δηλαδή ε, να μπουν στην ίδια γραμμή στον ίδιο κορβανά, αν θέλετε, οι χώρες που είναι στο ευρώ με τις χώρες που δεν είναι στο ευρώ όσον αφορά στη δυνατότητα αμφότερων να επιζητούν και να λαμβάνουν οικονομική βοήθεια. Νομίζω ότι ή του ευρώ μπορούν να τα καταφέρουν μόνοι τους, ωστόσο σε αυτή την οικονομική αναταραχή που επικρατεί παντού είναι σημαντικό το εργαλείο αυτό για τις χώρες που δεν έχουν το ευρώ. Η κυβέρνηση στη χώρα μου και φίλοι μου που βρίσκονται στην κυβέρνηση έχουν την αίσθηση ότι ε, μία Ιρλανδία π.χ. στην Ευρώπη θα προστατεύεται πάντοτε ε, και δεν θα έχει πότε πρόβλημα παρά τις αναταραχές. Αυτό είναι εσφαλμένο. Η δεκαετία ε, του 90 μας δίδαξε ότι κανείς δεν είναι προστατευμένος όταν έρχεται το τσουνάμι της κρίσης. Εξού και είναι αδύρυτη ανάγκη η ενίσχυση του συντονισμού. Και αυτό φαίνεται και με τις άλλες εκθέσεις που έχει συντάξει η Επιτροπή μας. Οφείλουμε αυτό να το κάνουμε και να καταλήξουμε σε ένα σύγχρονο χρηματοδοτικό εργαλείο και ευέλικτο. Και νομίζω ότι βεβαίως πρέπει να βελτιώσουμε και τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Και στη δική μας Επιτροπή και στο σύνολο του Κοινοβουλίου. Συμφωνώ λοιπόν με τη θέσπιση αυτών των νέων γραμμών πίστοσης, των δύο γραμμών πίστοσης και τον ρόλο του Κοινοβουλίου, των Εποπτικών Αρχών και της Ευρωπαϊκής ε, Κεντρικής Τράπεζας. Ίσως ένα στοιχείο λείπει, ένας κρίκος της αλυσίδας λείπει. Ο, η πρόταση κανονισμού ε, θέτει στο περιθώριο το ρόλο του Κοινοβουλίου ως προς τον προϋπολογισμό. Δηλαδή η Επιτροπή θα δανειστεί χρήματα από τις κεφαλαίες αγορές ε, τα οποία χρήματα θα εγγυώνται από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, που θα λειτουργήσει ως εχέγγυο. Ε, όμως το Κοινοβούλιο δεν θα έχει λόγο ως προς τις συνθήκες υπό τις οποίες θα δίδονται τα χρήματα αυτά στα κράτη-μέλη. Και αν κάποια χώρα δεν μπορεί να αποπληρώσει τα δάνεια τη, τότε ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα πρέπει να καλύψει το κόστος αυτό. Και άρα θα απαιτηθεί αύξηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και άρα αύξηση στη συνεισφορά των κρατών μελών στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Θα πρέπει αυτό να το σκεφτούμε περισσότερο και θα πρέπει να απαντηθούν δύο ερωτήματα. Πρώτον, η εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην έγκριση δανείων και γραμμών πίστοσης. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να έχει ένα ρόλο εποπτείας του προπολογισμού ως προς τη χρηματοδότηση των διαδικασιών και ως προς την εκταμίευση των διαφόρων δόσεων. Και δεύτερον, ποιε θα είναι οι επιπτώσει στον προπολογισμό των κρατών μελών. Πρέπει να εξετάσουμε αυτά τα δύο ερωτήματα στην έκθεση, στη γνωμοδότηση και ελπίζω οι εισηγητές να ε, καταλήξουν σε επαρκείς απαντήσεις. Κατά τα λοιπά, συμμερίζομαι απολύτως τις απόψεις της εισηγήτριας. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλά χέρια από τη στιγμή που η υπεύθυνη εισηγήτρια είναι η κυρία Ντανούτα Χιούμπνερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Σβέν, εξ ονόματος των Πρασίνων. Ναι, να ζητήσω συγγνώμη γιατί η σκιώδης εισηγήτρια Εύα Ζολή δεν είναι εδώ μαζί μας. Είχε συμμετάσχει πολύ δραστήρια ως προς την επίλυση της κρίσης στην Ισλανδία και ήταν ανώτατη σύμβουλος της κυβέρνησης εκείνη την εποχή. Διαγράφονται λοιπόν πολλές ομοιότητες ακόμα και σε χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω να μπορέσουμε όλοι να αντλήσουμε τα διδάγματα της σοφίας που απέκτησε από την παραμονή της στην Ισλανδία. Κατά τα λοιπά να ευχαριστήσω την κυρία Χιούμπνερ διότι έχει οργανώσει συναντήσεις με τους σκιώδες εισηγητές και ελπίζουμε πράγματι ότι αυτό το επικοδομητικό πνεύμα συνεργασίας θα συνεχιστεί. Ε, καταλαβαίνουμε και τη στηρίζουμε στην βούλησή της να συμπεριλάβει τα επιτεύγματα ε, που έχουμε εμείς πετύχει με την έκθεση «Κοζές». Υπ' αυτή την έννοια πολλές από τις ανησυχίες που είχαμε ήδη απεικονίζονται ε, στη, ε, στο τρέχον ε, κείμενο. Δηλαδή, κοινωνική δικαιοσύνη, στις συνθήκες ρεσιμότητας, δημοκρατικός έλεγχος για τα διάφορα προγράμματα. Αυτά όλα υπάρχουν. Και είναι καλό να αξιοποιήσουμε αυτή τη χρονική συγκυρία ώστε να κοιτάξουμε με ειλικρίνεια την κατάσταση των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης που έχουν λάβει διάφορα από αυτά τα κονδύλια. Ορισμένες χώρες θεωρούνται ως οι καλοί μαθητές στην κρίση του ευρώ. Ενώ συνάμα ε, τίνουμε να λησμονούμε την ε, οδύνη των ανθρώπων η οποία συνόδευσε τη σταθεροποίηση της μακροοικονομικής κατάστασης. Πάρα πολλοί άνθρωποι αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους αντιμετωπίζοντας το φάσμα της αυξανόμενης ανεργίας και της φτώχειας. Θα πρέπει λοιπόν με κάθε ειλικρίνεια να εξετάσουμε την κατάσταση σε κάθε μία από τις χώρες αυτές και να δούμε και τις κοινωνικές επιπτώσεις των διαφόρων προγραμμάτων που εφαρμόζονται πέρα από την οικονομική ανάλυση του εκάστοτε προγράμματος. Στη συνέχεια, εξίσου σημαντικό είναι να εξετάσουμε και τη διαδικαστική πλευρά της έκθεσης αυτής. Όπως είπατε και εσείς, κυρία Πρόεδρε, όλα αυτά γίνονται επί τη βάση του άρθρου 352 ε, και προβλέπονται ε, οι εξής ε, κανόνες. Εξετάζουμε έκθεση πρώτα ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ως αντίβαρο σε αυτό που κάνει η Επιτροπή και το Συμβούλιο. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα κατά τη γνώμη μου. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο ε, θα λάβουν πλήρως υπόψη τις επιθυμίες μας. Ίσως θα πρέπει να τους δοθεί ο λόγος για να μας απαντήσουν επ' αυτού και θα πρέπει και να εξετάσουμε και το δικό μας ε, εσωτερικό κανονισμό. Ε, πώς αντιμετωπίζουμε δηλαδή το θέμα αυτό. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις που βασίζονται στο άρθρο 352. Ε, όσο περισσότερο φτάνουμε στα όρια της συνθήκης, τόσο πιο δύσκολο αποδεικνύεται να αλλάξει η συνθήκη και όσο πιο δύσκολο αποδεικνύεται να αλλάξει η συνθήκη, τόσο περισσότερες προτάσεις θα δεχόμαστε με νομική βάση το άρθρο 352 όπου η θέση μας δεν είναι και ισχυρότερη. Ίσως η συγγήτρια ε, θέλει να συμπεριλάβει αυτό με το, ε, αυτή την έννοια του fiscal backstop και για τις χώρες που δεν είναι στο ευρώ. Είναι πολύ χρήσιμη πράγματι αυτή η συζήτηση ο ίδιος χρηματοδοτικός μηχανισμός που έχουμε χρησιμοποιήσει στην κρίση για να σταθεροποιήσουμε κυβερνήσεις θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ώστε να χρησιμεύσει ως backstop για την άμεση ανακεφαλοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Ε, δεν υπάρχει νομικό εμπόδιο κατά τη δική μας άποψη, ε, άρα θα μπορούσε κανείς να αναπτύξει περαιτέρω την εμπειρία που έχουμε με την εφαρμογή των διαφόρων μνημονίων και προγραμμάτων. Και τέλος, Νομίζω ότι ο δημοκρατικός έλεγχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, για το τι συμβαίνει στην κάθε χώρα που έχει μπει σε μνημόνιο είναι βασική μας ανησυχία και μέλημα. Αυτό το έχουμε αναφέρει στην έκθεση Κοζές και με το φόρτο εργασιών που έχει η δική μας Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, ίσως δεν έχουμε κάνει όσα πρέπει ε, για να εξετάσουμε σε βάθος τι τελικά συνέβη και σε ποιο βάθος συνέβη ε, στη Ρουμανία, στη Λετωνία και στις άλλες χώρες. Ναι, στείλαμε κάποιες αποστολές εκεί, αλλά δεν ε, δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή. Κάποια από τα προβλήματα που αντιμετώπισαν ήταν άμεσος απότοκος της κρίσης του ευρώ σε συνδυασμό πάντοτε με τοπικούς παράγοντες. Αυτό είναι αληθές. Η έκθεση όμως θα μπορούσε να τα αναφέρει αυτά, θα μπορούσε να εξετάσει ε, περαιτέρω ε, και τι θέλουμε εμείς ως Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων να κάνουμε για όλα αυτά. Ε, για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την συνεργασία της. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει πρόσωπο τη Ενωμένης ΕΕ, Αριστερά ή των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών εδώ. Θέλει κάποιο άλλο το λόγο. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια. Είχαμε, είχαμε τρεις ε, στόχους. Πρώτον, να ενισχύσουμε το δίχτυ ασφαλείας, εξυγχρονίζοντας το κείμενο και βάζοντας μέσα και την πρόοδο που έχουμε στα firewalls για ε, μεγαλύτερη ευελιξία στις, ε, στους δανεισμούς δεύτερον να βελτιώσουμε την εποπτεία και για μετά το πρόγραμμα. Και τρίτος στόχος, αλλά σημαντικός επίσης, ήταν η απλούστευση της γραφειοκρατίας για τις χώρες που εντάσσονται στο πρόγραμμα, όπως έχουμε και σε άλλα κείμενα. Έγινε δεκτή η πρόταση τον Ιούλιο, δηλαδή πριν να εγκύψει το Κοινοβούλιο στις προτάσεις Γκοζές. Είμαστε λοιπόν δεσμευμένοι σε μια προσπάθεια εξασφάλισης του ότι οι τροπολογίες που έχει καταθέσει το Κοινοβούλιο στην έκθεση Γκοζές και αυτές θα ενσωματωθούν στο κείμενο, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα εγκριθεί η δέσμη των δύο μέτρων, το two-pack, κάτι το οποίο για μας είναι βέβαια σημαντικό. Και όσον αφορά την ανακεφαλαιοποίηση, πρέπει να τονίσω, όπως είπε και ο εισηγητής σας, η εισηγητία σας μάλλον, ότι έχουμε κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά να χρησιμοποιήσουμε ε, το εργαλείο της άμεσης ανακεφαλαιοποίησης. Όχι νομικό πρόβλημα, είναι περισσότερο πρόβλημα οικονομικής ε, φύσεως, γιατί όταν κάνουμε επενδύσεις σε μετοχές equity investment είναι περισσότερο επικίνδυνο παρά όταν αγοράζουμε ομόλογα κρατικών δανείων. Γι' αυτό εγώ επειδή έχω αναλάβει το, την προετοιμασία στον ESM αυτού του εργαλείου υπάρχει μεγαλύτερος ε, κίνδυνος και ε, βέβαια να αντιδράσουν και οι οίκοι πιστοληπτικής ικανότητας. Ο κ. Σμιτ σωστά είπε για το backstop, το οποίο είναι σημαντικό για, το, για την αγορά των, του υπόλοιπου των μετοχών που δεν έχουν καλυφθεί δηλαδή από την εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Είναι ενδεχόμενο να υπάρξει αρνητική αντίδραση των οίκων πιστοληπτικής ικανότητας και αυτό να οδηγήσει σε υποβάθμιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτό εάν διατηρήσουμε σε χαμηλά επίπεδα τη χρήση του εργαλείου αυτού. Γιατί θεωρούμε ότι είναι δύσκολο μέσα στα παρόντα πλαίσια, αν και είμαστε έτοιμοι να διαρευνήσουμε και άλλες δυνατότητες με την εισηγήτριά σας. Υπάρχει ένα ακόμα εργαλείο το οποίο περιλαμβάνεται στον σταθεροποιητικό μηχανισμό, δηλαδή δάνεια προς τις τράπεζες για ανακεφαλαιοποίησή τους αυτό παρουσιάζει λιγότερα προβλήματα σε ό,τι αφορά τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο. Έχουμε συναντηθεί ήδη με τους συζητητές σας και είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε σε περαιτέρω συνεργασία και να συνεργαστούμε με, την, με το Κοινοβούλιο παρόλο που δεν είναι απόλυτα στο πλαίσιο της συναπόφασης. Θέλουμε όμως να συνεχίσουμε την καλή συνεργασία που έχουμε και στα άλλα κείμενα και σε αυτό. Έχω μία ερώτηση. Αν υπάρχει αρκετό χρόνος. Μου φάνηκε ενδιαφέρον αυτό που είπατε. Δύο ερωτήσεις. Αν καταλαβαίνω καλά, αυτό που γίνεται τώρα με το σταθεροποιητικό μηχανισμό είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια νομικού διαχωρισμού των δύο κινδύνων. Αυτό ίσως αποτελεί μια επιλογή και εν προκειμένου. Δηλαδή, αν δημιουργήσετε δύο διαφορετικές οντότητες, ίσως μπορέσετε να αποφύγετε το ενδεχόμενο μόλυνσης από το πιο επικίνδυνο τμήμα στο λιγότερο επικίνδυνο τμήμα. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι το επιχείρημα αυτό είναι ισχυρό γιατί να μην το χρησιμοποιήσετε. Ίσως πολιτικά να μην α, ικανοποιεί όλους. Αλλά εάν μπείτε σε κοινό σύστημα εποπτείας τραπεζών θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό backstop, γιατί αλλιώ πάλι προκαλείται ανισότητα. Και ανησυχώ πολύ, διότι μπορεί να μην δημιουργήσουμε κατάλληλε συνθήκε εν τέλει για να συμμετάσχουν πολλοί σε ισότιμη βάση. Αν τίνετε λοιπόν προ κάποια αρνητική κρίση, ποια είναι η εναλλακτική σα επιλογή. Και δεύτερο, μπορείτε να προβλέψετε νομικό διαχωρισμό των δύο. Και το δεύτερο, θα ήθελα να γνωρίζω τι εννοείτε όταν είπατε ότι θα λάβετε υπόψη σας την εργασία μας εάν εγκριθεί το λεγόμενο two-pack. Αυτός ο όρος είναι αρκετά ασυνήθιστος που βάζετε και διαρωτώ με εάν μπορούμε να βάλουμε όρους επί όρων επί όρων. Μπορείτε βέβαια να εννοήσετε ότι και το Κοινοβούλιο χρησιμοποιεί ανάλογες μεθόδους αλλά ίσως είναι καλύτερα να επανέλθουμε στο πνεύμα της ε, συνεργασίας. Ας αρχίσω από το τελευταίο σας ε, για να αποφευθούν οι εισδήποτε παρανοήσεις. Πολλοί από τους παρισταμένους εδώ έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά για το Tupac και θα είμαστε πολύ απογοητευμένοι αν αυτή η προσπάθεια αποβεί εισμάτιν. Με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να ερμηνεύσετε αυτό που είπα. Η Κομισιόν επίσης θα έχει και τη μεγαλύτερη, θα είναι πιο εύκολο δηλαδή να πλασάρει εντό εισαγωγικών, αν με επιτρέπετε, τι τροπολογίε του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, εφόσον το κείμενο αυτό θα έχει φτάσει σε νομική οριμότητα. Έρχομαι τώρα στην πιο τεχνική σα ερώτηση. χωρί να θέλω να προκαταλάβω με οποιοδήποτε τρόπο το γεγονό ότι θα υποστηρίξουμε την ενσωμάτωση των τροπολογιών σα στο κείμενο, επαναλαμβάνω, θα τι υποστηρίξουμε, κύριε Γκίγκολτ, μην με παρανοήσετε. Προσπαθούμε λοιπόν μέσα στο ESM να βρούμε τρόπο νομικού διαχωρισμού. Για παράδειγμα με τη δημιουργία του SPV. Εν προκειμένου δεν έχουμε βρει ακόμα τρόπο να το πράξουμε χωρίς πολύ αρνητική ε, επίπτωση στη δανειολητική ικανότητα. Εξακολουθούμε να το συζητούμε αυτό με τους συναδέλφους του ESM, αλλά τεχνικά είναι δύσκολο. Η οίκη επιστολιπτικής ικανότητας, ακόμα και για default σχεδόν στο 1, στη μονάδα, θεωρούν ότι έχει πολύ αρνητική επίπτωση. Θέλουμε να αποφύγουμε λοιπόν παρόμοια επίπτωση στον μηχανισμό ισοζυγίου πληρωμών, εκτός αν βρούμε ένα μαγικό ραβδάκι για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να αναλάβουμε σημαντικό κίνδυνο, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Θέσατε επίσης το ερώτημα των backstops για τον μηχανισμό εποπτείας και αυτό βέβαια είναι κέριο θέμα. Για τις χώρες που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν και που αναμένω να καλυφθούν από το μελλοντικό Ταμείο Εκαθάρισης Τραπεζών, το οποίο θα δημιουργηθεί στα επόμενα χρόνια, χρειάζεται ένα backstop. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο σταθεροποιητικός μηχανισμός από μόνος του, γιατί αυτός εκτείνεται μόνο στις χώρες ζώνης ευρώ. Θα αναζητήσουμε λοιπόν και άλλες δυνατότητες. Για παράδειγμα, μαζί με την γραμμή πίστοσης του ESM μπορεί να έχουμε και γραμμή πίστοσης από την ίδια την ενδιαφερόμενη χώρα. Αλλά είμαστε ανοιχτοί και σε άλλες προτάσεις βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή του προβληματισμού μας. Ντανούτα, ευχαριστώ όλες και όλους. Ελπίζω ότι η έκθεση θα είναι ιδιαίτερα πλούσια στο τέλος. Είναι και η στιγμή που μπορούμε να σκεφτούμε πράγματα τα οποία μπορούν να εμπνεύσουν και τα άλλα θεσμικά όργανα για το μέλλον όχι απαραίτητα μόνο να ε, βρούμε συγκεκριμένες λύσεις τώρα. Πολύ σύντομα τώρα για αυτά τα fiscal backstop της για το Ταμείο τη Εκαθάριση που για την ώρα θα οργανωθεί εθνικά. Στο το αφήσουμε λοιπόν λίγο στην άκρη. Αλλά για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και το backstop που είναι απαραίτητο εκεί. Το θέμα αυτό παραμένει ακόμα κρίσιμο. Διότι ακόμα αντιμετωπίζουμε πολλούς κινδύνους στον τραπεζικό τομέα και ιδίως μετά από την εισαγωγή του εποπτικού μηχανισμού στις χώρες οι οποίες λειτουργούν με θυγατρικές τραπεζών, εκεί υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα όταν θα υπάρχουν δύο κατηγορίες του τραπεζικού τομέα, δηλαδή ο ένας θα εποπτεύεται από ένα σημαντικό όργανο με καλή φήμη στην Ευρώπη και μια κατηγορία της αγοράς η οποία δεν θα τελεί υπό την εποπτεία. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος και γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε από την αρχή ποια πράγματα μπορεί να συμβούν στο μέλλον. Και γι' αυτό κατανοώ ότι το θέμα αυτό των ενδεχόμενων αλλαγών στη συνθήκη του ESM και συμμετοχή με κεφάλαιο των συμμετεχουσών χωρών που θα τους επιτρέπεται μετά να χρησιμοποιήσουν αυτήν αυτό το backstop για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι μια δυνατότητα που εξακολουθεί να υπάρχει δύσκολη βέβαια νομικά γιατί είναι και οδυνηρή διαδικασία. Καταλαβαίνω βέβαια και η δεύτερη επιλογή που είναι αυτή η διευκόλυνση αλλά εδώ έχουμε το πρόβλημα της χρηματοδότησης που είναι πραγματικό πρόβλημα και θα το αντιμετωπίσουμε κατά πάσα πιθανότητα αν δείτε από πού μπορούν να προέλθουν τα χρήματα. Αλλά υπάρχει και η τρίτη δυνατότητα ανάμειξης του κεφαλαίου με συμμετοχή και κεφαλαίων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. για να κινηθούμε προς μια επιλεγμένη κατεύθυνση, όμως να μην αφήσουμε την κατάσταση χωρίς καμία λύση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Γι' αυτό και εργάζομαι πάνω σε αυτή την πρόταση, εξετάζω αν είναι δυνατόν να γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Ένα όργανο δύο επιπέδων, ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση του κοινοτικού προϋπολογισμού. Μπορεί να είναι και αυτό μια επιλογή. Αλλά ας μην μπούμε βαθύτερα στη συζήτηση. Θα ευχαριστήσω όλες και όλους για τη συνεργασία μέχρι τώρα στο φάκελο αυτό και προς την πρόεδρό μας. Μπορούμε να κάνουμε παν το δυνατόν, ξέρω πόσο δύσκολο είναι βέβαια, για την έκθεση ένι, που νομίζω ότι και αυτό θα είναι καλή λύση. Thank you uh, Η πρόεδρος Μπόλου, ευχαριστώ. θα πρέπει να υποβληθεί στην επόμενη διάσκεψη των ε, Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για να λάβουμε την έγκρισή τους το δυνατόν συντομότερο. Εγώ προτείνω να αρχίσετε την σύνταξη του εγγράφου και εάν θα καταλέξει ως έννοι ή ως ψήφισμα αυτό θα το δούμε. Θα το συζητήσουμε και με τους συντονιστές, τις επιπτώσεις δηλαδή, απέναντι και στις άλλες εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλία. Δεν μπορώ να σας απαντήσω λοιπόν αυτή τη στιγμή, αλλά το εξετάζουμε. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα ακόμη, αλλά επειδή έχουν αρχίσει επειδή έχουν αρχίσει ήδη οι ισχυοδησηγητές. Ελπίζω να μπορέσετε να προχωρήσετε και να έχετε κάτι έντιμο σύντομα. Είναι βέβαια κάπως ασαφή αυτά που σας προτείνω, αλλά βρισκόμαστε και κάτω από δύσκολες συνθήκες, διότι μεταξύ άλλων είναι και μεγάλος όγκος εργασίας και υπάρχουν και πολλές διαφορετικές εκθέσεις ε, πρωτοβουλίας. Θα προχωρήσουμε τώρα στο υπαριθμό 7 διακανονισμό αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κεντρικά αποθετήρια. Είμαστε σχεδόν α, ακριβώς μέσα στον χρόνο που είχαμε προβλέψει, 9 και 40 είχαμε πει, αν και ενδεικτικά βέβαια, θα εξετάσουμε τις τροπολογίες και θα δώσω τον λόγο στο, στην εισηγήτρια Κέι Σουίνμπερν Έχουμε κάνει συναντήσεις σκιωδών και ε, συνεργατών τους και έχω υποβάλει ένα συμβαστικό κείμενο κυρίως τεχνικών τροπολογιών και έχω επίσης διανύμει και την ενδεχόμενη βάση για μια διακαμπατική συμφωνία για το ΣΥΣΤΗ με τραπεζικές άδειες για να επιτρέψουμε να μπουν και νέες ε, τράπεζες στην αγορά. Το κείμενο λοιπόν ε, κυκλοφορεί και οι σκιώδεις συγκητές ελπίζω ότι το εξετάζουν για να δουν εάν ικανοποιεί όλες τις πολιτικές ομάδες. Ίσως σήμερα πολλοί από τους σκιώδεις συγκητές θα θέλουν να συζητήσουν αυτό το κείμενο, μιας και το αρχίσαμε την προηγούμενη ε, εβδομάδα στο Στρασβούργο. Προτιμώ με την ευκαιρία αυτή να ακούσω τις απόψεις των σκιωδών εισηγητών, μιας και έγινε η προκαταρκτή ή μάλλον ας πούμε η πρώτη συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Τότε λοιπόν θα προχωρήσω αμέσως στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τον Herbert Dorfman. Μην λησμονείτε ότι Η συνεδρίασή μας μεταδίδεται από το διαδίκτυο και οι άνθρωποι που ενδεχομένω παρακολουθούν δεν γνωρίζουν το περιεχόμενο των κειμένων. Ο κ. Ντόρφμαν. Πράγματι, η συζήτηση στρέφεται γύρω από το άρθρο 52. Δηλαδή το ερώτημα ποια μορφή θα λάβουν οι τραπεζικές υπηρεσίες των κεντρικών αποθετηρίων. Νομίζω, ή μάλλον ευχαριστώ την κυρία Σουίνμπερν, την βασική εισηγήτρια δηλαδή, για την πρόταση που κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα και που νομίζω ότι κατευθύνεται βασικά στη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω ότι πρέπει να καταλήξουμε σε μια ρύθμιση η οποία να προβλέπει χωρισμό μεταξύ τραπεζικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων των κεντρικών αποθετηρίων, όπου βέβαια θα πρέπει να προβλεφθεί και κάποια εξαίρεση. Όμως, η οποία θα πρέπει να περνά από μια σαφή ευρωπαϊκή διαδικασία εγκρίσεως. Θα πρέπει να υπάρχει διαδικασία εγκρίσεων ώστε τα κεντρικά αποθετήρια να μπορούν να παίξουν σε ένα πεδίο ισότιμου ανταγωνισμού σε όλη την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες μέλη όπου, η δραστηριότητα το, όπου θα, θα συντελείται η δραστηριότητα των κεντρικών αποθετηρίων θα πρέπει να υπάγονται αυτές οι δραστηριότητες στην ε, διαδικασία που περιέγραψα και η ΕΣΜΑ θα πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο. Μόνο τότε νομίζω ότι θα υπάρχει πραγματικά ανεξάρτητη διαχείριση όλων των κεντρικών αποθετών. Εφόσον η κεντρική η τα κεντρικά αποθετήρια αποφασίσουν να προσφέρουν στην αγορά ξεχωριστά μοντέλα, δηλαδή να δημιουργήσουν δική τους τράπεζα η οποία θα προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες, Νομίζω ότι θα είναι τότε λογικό αυτές οι τράπεζες να απαιτείται να διαθέτουν πλήρη άδεια εκτέλεσης τραπεζικών υπηρεσιών. Αλλιώς νομίζω δεν έχει πολύ νόημα. Μπορούμε όμως να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε μια πρόταση συμβιβαστική και νομίζω ότι στα όματα της πολιτικής μου ομάδας τουλάχιστον υπάρχει δυνατότητα να ε, συνταχθεί μια, να βρεθεί μια λύση την οποία να υποστηρίξουμε. Τώρα για το υπόλοιπο, γιατί δεν υπάρχει βέβαια μόνο το άρθρο 52, έχουμε και έναν αριθμό τροπολογιών με την πρόθεση να διασφαλιστεί ένα σκανδιναβικό μοντέλο των κεντρικών αποθετηρίων, διότι στις χώρες αυτές υφίσταται ένα συγκεκριμένο μοντέλο με το οποίο εργάζονται οι κεντρική αποθέτηση και θα πρέπει να βασιστούμε σε αυτό, διότι αφενός δεν περιλαμβάνει κινδύνους, αφετέρου προσφέρει επαρκή διαφάνεια. Υπάρχουν λοιπόν τροπολογίες που κατευθύνονται προς τα εκεί, από την δική μας επίσης πολιτική ομάδα ή που υποστηρίζονται από αυτήν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους συνδέσμους, links, μεταξύ των κεντρικών αποθετηρίων των διαφόρων χωρών μελών, νομίζουμε ότι δεν είναι λογικό, όπως προτείνει η Κομισιόν, όλοι οι σύνδεσμοι, όλα τα links που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των κεντρικών αποθετηρίων μεταξύ χωρών μελών, να εγκριθούν όλα αυτά δηλαδή, θα πρέπει να εγκρίνονται τα links αυτά μόνο εφόσον είναι διαλειτουργικά. Δηλαδή, θα πρέπει όλα, όλες οι απλές διασυνθέσεις, τα απλά links δηλαδή, να εξαιρούνται από την διαδικασία εγκρίσεων. Ευχαριστώ. Um, thank uh, Σας ευχαριστώ. Τώρα για την S&D. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το επικοδομητικό πνεύμα συνεργασίας της. Έχει υποβάλει ήδη μια πρώτη ένα πρώτο γύρο προτάσεων ε, συμβιβαστικών λύσεων και εγώ είμαι διατεθειμένος να συνεργαστώ πλήρως και μάλιστα με επικοδομητικό τρόπο για την επίτευξη συμφωνίας. Όλες αυτές οι τροπολογίες που παρουσίασα θέλω θέλουμε να έχουμε σκοπό να ενισχυθούν τα κεντρικά αποθετηρία τίτλων και να είναι πραγματική υποδομή της αγοράς αυτής. Να υπάρχει νομική ασφάλεια, ένα ασφαλές πλαίσιο, διαφανές, αποτελεσματικό και με σαφήνεια να διευκρινιστεί αυτό το οποίο είναι απαραίτητες υπηρεσίες και αυτό το οποίο είναι επικουρικές υπηρεσίες. Και πρέπει να το συζητήσουμε αυτό αν είναι απαραίτητη η υπηρεσία των ε, κεντρικών αποθετηρίων τίτλων και πρέπει να το έχουν οι τράπεζες ή άμα είναι επικουρικές υπηρεσίες. Εάν είναι επικουρικές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι διαφορετικοί οι η μεν και η δε για να μην υπάρξει μόλυνση, μετάδοση και εξάπλωση μάλλον ε, των προβλημάτων. Και θα πρέπει να δίδεται επαρκές χρονικό διάστημα ώστε οι φορείς, ε, οι εμπλεκόμενοι να ε, προσαρμοστούν και να, και να παρουσιάσουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Όλα αυτά είναι στη, στη γραμμή που προτείνουμε. Ε, και νομίζω ότι έτσι θα καταφέρουμε να έχουμε συμβαστικές λύσεις. Θέλουμε να εγγυηθούμε τη θέση και τα δικαιώματα ε, των μετόχων αλλά και των επενδυτών γιατί είναι μια υποδομή της αγοράς και θα πρέπει στο έσμα να υπάρχουν ε, τα τεχνικά ε, πρότυπα και να Υπάρχει και η προοπτική του Target 2 Securities, αυτή η πλατφόρμα για τον διακανονισμό αξιογράφων στην Ευρώπη. Να γίνονται όλα δηλαδή με τυποποιημένα πρότυπα για να έχουμε ανοιχτές διαδικασίες και να μην γίνονται διακρίσεις κατά την ε, ρευστοποίηση και να υπάρχει και ευελιξία ως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και να προβλέπονται και οι απαιτήσει της Βασιλείας ε, για το όσο το πιο σύντομο χρονικό διάστημα για τις προθεσμίες. Στο Στρασβούργο είχαμε μια πρώτη επαφή με πολύ θετικό πνεύμα και ελπίζουμε ότι θα ε, προχωρήσουμε για να έχουμε μια ικανοποιητική συμφωνία για όλους. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι σκιώδης, για την Άλντε και μου δίνω λοιπόν το λόγο ως σκιώδης της ε, Άλντε υπό αυτή μου την ιδιότητα. Στην ομάδα μου οι απόψεις διαφέρουν, όπως νομίζω οποτεδήποτε εξετάζει κανείς κάποια από αυτά τα θέματα. Κάθε φορά που το βλέπει κανείς μπορεί να αλλάξει τη γνώμη του. Αλλά Εν γέννη αποφασίσαμε πως η εξαίρεση, η προσέγγιση μάλλον εξαίρεσης από πλευρά της ε, Κομισιόν για την απέτηση από τα κεντρικά αποθετήρια να διαχωρίσουν τις τραπεζικές τους υπηρεσίες από τις υπόλοιπες ε, δεν ήταν η σωστή προσέγγιση και γι' αυτό τη διαγράψαμε και εξετάζοντας το κατά πόσο θα πρέπει να ε, διαχωριστούν τα κεντρικά αποθετήρια με τραπεζικές άδειες, τα διεθνή δηλαδή αποθετήρια, από την προοπτική του κινδύνου που θα πρέπει δηλαδή κανείς να σκεφτεί πως αυτός είναι ένας τρόπος για να μειωθεί ο κίνδυνος, εγώ νομίζω πως θα πρέπει να γίνει περισσότερη εξολόγηση και προετοιμασία εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Ε, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να έχουμε υπόψη μας, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει έχει πια λυθεί. Εν πάση περιπτώσει, για τα κεντρικά αποθετήρια τα οποία θα συνεχίσουν να ασκούν τραπεζικές δραστηριότητες αλλά και καθαριστικές, θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ αυστηροί και να αποδείξουμε στις αρμόδιες αρχές ότι εάν κάποιο αποθετήριο συναντήσει δυσκολίες, οι τραπεζικές του δραστηριότητες θα συνεχίσουν ε, κανονικά. Ε, και οι απαιτήσει ε, πρόνοιας, θα υπάρχουν στο άρθρο 4 να είναι στεναρές, να υπάρχουν δηλαδή προγράμματα ανάκτησης και εκαθάρισης που θα συμμορφούνται προς την οδηγία για τη διαχείριση της κρίσης. Θα δημοσιεύεται δηλαδή λεπτομερής ανάλυση για τις ενδοημερήσιες ρευστότητες και τους κινδύνους ρευστότητα, ε, όπως προβλέπεται από την οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Έχουμε εξάλλου οι ρυθμίσεις 1 και 2 ε, ε, μπορεί να είναι αντιανταγωνιστικές αν δούμε δηλαδή το τι ισχύει για τα κεντρικά αποθετηρία. Πολλοί άνθρωποι δηλαδή στην ουσία έχουν βάλει το χέρι ήδη στη φωτιά με τον έναν τον άλλο τρόπο και δεν, είναι αυτό, δεν σημαίνει ότι απαραίτητο θα βρούμε καλύτερη κατάσταση. Αυτό που με ενδιαφέρει ωστόσο είναι να αναζητήσουμε συμμετρικές ρυθμίσεις όπου το αποθετήριο στην ουσία είναι μια περιορισμένη τράπεζα. Ίσως αυτό να είναι κάπως θεωρητικό, αλλά εν πάση περιπτώσει προς αυτού του είδους τις συμμετρικές αντιστοιχίες θα πρέπει να τίνουμε, γιατί να μην έχουμε διακρίσεις, να μην είναι μονόδρομες οι καταστάσεις, αλλά αμφίδρομες, εφόσον δεν θέλουμε να υπάρχουν διακρίσεις. Πιστεύω πως η διαφάνεια θα βοηθήσει πολύ. Να πω και δύο πράγματα για το άρθρο 7 και την ε, πειθαρχία ε, ε, διακανονισμού. Είναι σημαντικό αυτό στην ε, ο καθεστώς και υπάρχουν ε, μη θελημένες συνέπειες στις αγορές ολόκληρη την Ένωση. Το τελευταίο που θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε αντικίνητρα για τις μικρομεσαίες να χρησιμοποιούν τις κεφαλαϊκές αγορές, τις αγορές κεφαλαίου, γιατί υπάρχει περιβολικός κίνδυνος για τους επενδυτές όταν αγοράζουν τα αξιογραφά τους. Αυτό ήταν πολύ άσχημο, το να αποθαρρυνθούν δηλαδή οι μικρομεσαίες από το να πάνε στις κεφαλαγορές από τη στιγμή που υπάρχουν προβλήματα στο δανεισμό και από τις τράπεζες. Οι μικρομεσαίες ε, λοιπόν και οι λιγότερο ρευστείς ε, μετοχές θα πρέπει να μην καλύπτονται. Αυτό θα μπορούσε να είναι στη διακριτικότητα των αρμοδίων αρχών. Υπάρχουν κάποιοι έλεγχοι που δεν είναι για όλους, αλλά πρέπει να μπορέσουμε να διατηρήσουμε ρευστότητα. Ενώ είναι αλήθεια πως ε, τα αξιόγραφα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ε, τα διάφορα είδη ρευστότητα που ανέφερα βρίσκονται σε διάφορα στάδια της, ε, του κύκλου ζωής τους, θα πρέπει ωστόσο να παραμείνουν ελκυστικά για τους επενδυτές αυτά τα δύο αξιόγραφα. Να είμαστε ρεαλιστές για τις αγορές που υπάρχουν ε, και δεν θέλουμε να αναγκάσουμε, να διώξουμε τον κόσμο από τις διαφανείς αγορές προς τις λιγότερο διαφανείς λύσεις. Έχω την εντύπωση λοιπόν πως είναι λογικό να δώσουμε στήριξη για ένα από αυτά τα καθεστώτα και να την αρνηθούμε στα υπόλοιπα. Επιμένω λοιπόν να κάνουμε κάτι για τα λιγότερα ρευστά μέσα. Πέρα λοιπόν από αυτές τις ρυθμίσεις πρόσβασης για 44α και 52α, ο κανονισμός ολοκληρώνει τις ρυθμίσεις πρόσβασης για το ΕΜΙΡ ε, και είναι πολύ σημαντικό οι δύο οδηγίες για την ανακεφαλαιοποίηση αλλά και για τα κεντρικά αποθετήρια να μην χρησιμοποιούνται ε, ως στρέβλωση στην αγορά. Δεν μπορούμε να έχουμε υποδομέ που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην νέα αγορά. Γιατί αν το πράξουμε αυτό, τότε θα δώσουμε λαβή για περισσότερες συστημικές υποδομές και δυνητικές εγγυήσεις των φορολογουμένων, πράγμα που οδηγεί στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θέλουμε. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, τότε χρειάζεται η Κομισιόν να παρέμβει ή να προβεί σε νέες νομοθετικές προτάσεις. Άρθρο 33 είναι λογικός ο τρόπος με τον οποίο παίζει ρόλο το κεντρικό αποθετήριο στις συναλλαγές δανεισμού αξιογράφων αν μπορούν οι πληροφορίες να δίνονται στις αρμόδιες αρχές, την EPA, την ESPA, την ΕΚΤ και το... την ESRB. Ξέρω πως αυτή τη στιγμή υπάρχει ε, μία δυνατότητα απόθεσης στην έκταλα, πληροφορίες πρέπει να είναι εύκολα διαθέσιμες. Και μετά από την την πρωτοβουλία του CFSP να δημιουργηθεί μια δυνατότητα αναγνώρισης, μια, ένα είδος ταυτότητας ε, έτσι ώστε να γνωρίζουμε τις συναλλαγές. Αυτό συμφωνεί με τις εργασίες τις οποίες ε, αναφέρθηκα. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε, και αυτό βρίσκεται στο άρθρο 2, τα κεντρικά αποθετήρια να χρησιμοποιούν διαδικασίες διεθνούς διαφάνειας ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα εμπόδια πρόσβασης για άλλους συμμετέχοντες υποδομές. Νομίζω ότι αυτά είχα να πω για την ώρα. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά του. Λυπάμαι που χρειάζεται να δουλέψω και εξ όταν ε, ε, χρειάζεται να συμμετέχω σε τον τριμερή διάλογο, αλλά τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή του Προέδρου. Λοιπόν, και τώρα εξ ονόματος των Πρασίνων, ο Ζαν Πολ Μπεσέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να πω στην κυρία Σουίνπερ, την εισηγήτριά μας, ότι χάρη στη δουλειά της ε, βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση για την επίτευξη ικανοποιητική συμφωνίας. Γενικώ συμφωνούμε με την έκθεση αυτή, εκτός από ένα σημείο το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί σε αυτό το στάδιο. Ομιλώ για το περιβόητο άρθρο 52 πώς ε, με τρόπο ευανάγνωστο, σαφή και αποτελεσματικό θα ξεχωριστούν οι τραπεζικές δραστηριότητες μέσα στον κανονισμό, ώστε να μην εξαπλώνονται οι κίνδυνοι του τραπεζικού συστήματος στα κεντρικά αποθετήρια τίτλων. Ποιο φράγμα θα υψωθεί ε, ώστε να αποφευθεί αυτή η πάντοτε πιθανή και πάντοτε καταστροφική εξάπλωση. Η κυρία Σουίνμπεργκ μας εξέφρασε την ε, θέλησή της να προτείνει ένα φράγμα ανυπέρβλητο, δηλαδή σαφή διαχωρισμό δραστηριοτήτων. Εξού και η σύμβαση που προτείνεται, η συμβαστική λύση που προτείνεται σε αυτό το στάδιο παραμένει κατά την άποψή μας σχετικά ασαφής και επιτρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να έχουμε κάποιες οντότητες μη διαχωρισμένες από τις άλλες που είναι ξεκάθαρα διαχωρισμένες και έτσι το σύστημα είναι διτό, περίπλοκο και μπορεί να υπόκειται να επιδέχεται ναι, ναι, να αποβεί προβληματικό και να υπάρξουν ανεπάρκειες και ελλείψεις. Δηλαδή να, δεν, είναι αδιαπέραστο το εμπόδιο και ο, ο διαχωρισμός. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε περιορισμένη τραπεζική άδεια στην περίπτωση ε, τράπεζας με δραστηριότητα περιορισμένη και διακεκριμένη, ξεχωριστή. Και θα μπορεί ο στόχος αυτός να ισχύσει για μια συγκεκριμένη μεταβατική περίοδο, δύο-τριών ετών. Και μπορούμε να προβλέψουμε και εξαίρεση ή παρέκκληση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ώστε να μπορέσει ο κλάδος να προσαρμοστεί στις νέες διατάξεις. Συνοπτικά, η θέση μας είναι πολύ απλή και τη συζητούμε με την κυρία Σουίνμπεργκ. Ε, θα τηρήσουμε απαρέγκλιτα την αρχή του διαχωρισμού και θα έχουμε ρεαλισμό και ευελιξία στην εφαρμογή της αρχής αυτής για το πρώτο ε, χρονικό διάστημα, ε, το μεταβατικό. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κάποιος από την Ενωμένη Ευρωπαϊκή Αριστερά. Η Μάριον Τίσεν θέλει το λόγο. Θέλει και κάποιος άλλος το λόγο. Πρώτα η Σάρα και μετά η Μάριον Τίσεν. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά της. Πράγματι, η ίδια αντιμετώπιση θα πρέπει να επιφυλάξουμε και στο μοντέλο της άμεσης διακράτησης και στο μοντέλο Omnibus Συμφωνώ με τον συνάδελφο που μίλησε για το ε, μοντέλο το σκανδιναβικό που είναι πιο διαφανές. Πρέπει να έχουμε τις καλύτερες δυνατές ρυθμίσεις. Προσπάθησα να είμαστε πιο φιλόδοξοι στις προτάσεις μας. Έχουμε τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο πληρωμών και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε και τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο αξιογράφων. Στην τροπολογία μου την 128 λέμε ότι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αγοράς για το διακανονισμό των αξιογράφων θα πρέπει να είναι ο στόχος ώστε να λειτουργεί σωστά η εσωτερική αγορά. Και αν αυτός είναι όντως ο στόχος μας, τότε πρέπει να υιοθετήσουμε κοινά πρότυπα και πλήρη διαλειτουργικότητα όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφούνται με τα ίδια κοινά πρότυπα όπως ισχύει και στον Ενίο ευρωπαϊκό χώρο πληρωμών και όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι διασυνδεδεμένοι ώστε να μπορούν να αγοράζουν και να πολλούν αξιόγραφα τόσο εύκολα όσο θα το έκαναν και στη δική τους χώρα. Και στην, στον τροπολογία μου την 131 αναφέρεται ότι θα πρέπει ένας επενδυτής να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και να μπορεί ε, κάποιος να επενδύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλα τα αξιόγραφα. Ε, προτείνεται από το 2017 ο διακανονισμός να μειωθεί σε μία εργάσιμη ημέρα μετά την συναλλαγή. Και μετά το 2020 ο διακανονισμός θα πρέπει ε, να γίνεται την ίδια ημέρα, σε πραγματικό χρόνο δηλαδή. Είναι ένας στόχος αυτός για το μέλλον βέβαια. Είμαι βέβαιη όμως ότι έτσι θα εξοικονομήσουμε πάρα πολλά χρήματα και θα επιτύχουμε ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια. Νομίζω ότι οι τροπολογίες μου προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται. Ευχαριστώ την εισηγήτρια και προσβλέπω σε επικοδομητική συνεργασία μαζί της. Ευχαριστούμε. Η Μάριαν παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι εξαιρετικά σύντομη. Στις τροπολογίες μου εστιάζομαι στη συγκεκριμένη ε, πτυχή, δηλαδή στον υποχρεωτικό διαχωρισμό των ε, τραπεζικών ιδρυμάτων και στο μοντέλο 2 συν 2. Σημερίζομαι την άποψή σας, κυρία Πρόεδρε, και ε, συμφωνώ τους με τα κίνητρα, με τις αιτίες για τις οποίες εκφράσατε εσείς τις επιφυλάξεις σας. εγώ δεν έχω συναντηθεί με κανέναν που να με έχει πείσει πραγματικά ότι το μοντέλο 2 συν 2 θα πρέπει να αποκτήσει υποχρεωτικό χαρακτήρα και να γίνει τελικά η μόνη μας δυνατότητα. Νομίζω ότι θα μπορούσε να επικρατήσει το μοντέλο 2 συν 2 και να έχουμε και το 1 συν 1. Ε, να συμβιώσουν αυτά τα δύο μοντέλα τα οποία θα υπόκεινται στους κανόνες τους προληπτικούς, που είναι και αυστηροί. Και έτσι θα μπορούσαν όλοι να οργανώσουν τις δραστηριότητές τους επί ίσης όρης, οι φορείς δηλαδή και οι εμπλεκόμενοι. Θεωρείτε ότι θα είναι λιγότερος ο κίνδυνος. Δεν είμαι σίγουρη. Συμφωνώ με το να υπάρχει μεγαλύτερη αρμοδιότητα. Συμφωνώ με το να υπάρχουν όσο το δυνατόν μικρότεροι και λιγότεροι κίνδυνοι. Θα τα επιτύχουμε όμως αυτά με αυτό που μας προτείνει η συγκήτρια, Αναρωτιέμαι και αμφιβάλλω. Και γι' αυτό έχω παρουσιάσει διάφορες τροπολογίες. Πιστεύω ότι τα δύο αυτά μοντέλα θα πρέπει να λειτουργήσουν παράλληλα και δεν θα πρέπει να ε, υποχρεώσουμε όλους να συμμορφούνται με το υποχρεωτικό μοντέλο 2 συν 2. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, Τζάνης από την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις γιατί δεν έχω ε, διαβάσει λεπτομερώς τις προτάσεις της κυρίας Σουίνπερκ. Θα βασιστώ μόνο σε όσα άκουσα εδώ σήμερα. Πρώτον, ως προς το διαχωρισμό των τραπεζικών υπηρεσιών από τις υπηρεσίες κεντρικών αποθετηρίων τίτλων. Δεν θα εκπλαγείτε, αλλά όπως είπαμε και στη δική μας πρόταση προέχει η ασφάλεια και αυτό το μοντέλο είναι και το πιο ασφαλές. Τώρα, ως προς τα σχόλια της κυρίας Τίσεν, ότι τα δύο ε, συστήματα θα πρέπει να λειτουργήσουν παράλληλα. Εμείς προτιμούμε το εξή σύστημα. Ε, το μοντέλο διαχωρισμού να είναι ο κανόνας και ε, να υπάρχουν και εξαιρέσεις, γιατί αυτό το μοντέλο είναι αυτό που προσφέρει ε, αθρηστικά πολλά πλεονεκτήματα. Τώρα, ως προς τα δικά σας σχόλια, κυρία Πρόεδρε, για την περίοδο συμμετοχής, buy-in, Καταλαβαίνουμε το πνεύμα των τροπολογιών των ε, σκιωδών εισηγητών, καταλαβαίνουμε την ανάγκη να υπάρχει ευελιξία για τα ζητήματα αυτά. Ωστόσο, η νομοθετική ρύθμιση πολύ συγκεκριμένων εξαιρέσεων πάντοτε θα είναι δύσκολη και πάντοτε είναι δύσκολο να δοθεί νομικός ορισμός αυτών των ε, εξαιρέσεων. Βέβαια μπορούμε να εξερευνήσουμε διάφορες δυνατότητες πώς μπορούμε να το ρυθμίσουμε το θέμα αυτό, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Μία επιλογή ενδεχομένως για να καθυστερήσει η, περιοδο η περίοδος buy-in για ε, συγκεκριμένα προϊόντα, επιλογή ε, του αντισυμβαλόμενου να ε, αποφασίσει αναπερίπτωση, π.χ. και Τώρα, ως προς το σκανδιναβικό μοντέλο, και το μοντέλο ε, διακράτησης τύπου Omnibus ή το μοντέλο διακράτησης άμεσης. Καλό είναι να σημειώσουμε το γεγονός ότι εξετάζουμε την νομοθεσία περί αξιογράφων αυτή τη στιγμή εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ίσως κάποια ζητήματα θα πρέπει να τα προσεγγίσουμε πιο οριζόντια να το εξετάσουμε αναπερίπτωση για να δούμε εάν σε κάθε περίπτωση αρμόζει περισσότερο η οριζόντια προσέγγιση. Και αυτό προγραμματίζεται το προσωπικό μας να το αναλάβει ως καθήκον την άνοιξη της επόμενης χρονιάς. Να το δω και να μην το πιστέψω, λέει η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Okay. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ όλους για τις παρατηρήσεις σας. Νομίζω πως όλοι οι συγητές και οι σκιώδεις έχουμε καταλάβει ότι ο συνδυασμός ε, αποθετηρίου και τράπεζας θα πρέπει να είναι εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Νομίζω πως όλοι συμφωνούμε ε, γι' αυτό. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτοί που τώρα λειτουργούν με το συνδυασμένο μοντέλο θα πρέπει να επιτραπεί να συνεχίσουν επαόριστον ή αν θα πρέπει να τους δώσουμε μια περίοδο μεταβατική για να διαλέξουν το ένα από τα δυο. Νομίζω αυτό θα μας, απασχολήσει κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων, μετά τα Χριστούγεννα, όχι κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Αλλά νομίζω πως είναι σημαντική συζήτηση, γιατί η Κομισιόν είναι πεπισμένη πως υπάρχουν πλονεκτήματα για το διαχωρισμό και άρα θα πρέπει να κάνουμε αυτή την εισβάθος συζήτηση, ώστε να δούμε αν θα μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο για να το ξεπεράσουμε. Ε, Επίσης πιστεύω πως όσον αφορά την πειθαρχία διακανονισμού, οι τροπολογίες που εγώ υπέβαλα στη δική μου έκθεση και η πρότασή μου είναι ε, προαιρετική. Είναι μετά από ζήτηση του δικαιούχου ε, όσον αφορά τις, ε, τη ρευστότητα, μάλλον τις λιγότερο ρευστές μετοχές αλλά νομίζω πως θα πρέπει να καλύψουμε την πλειοψηφία των ε, αξιογράφων και όχι την μειοψηφία ε, για το βασικό όγκο αξιογράφων στην, ε, σε ολόκληρη την Ένωση. Νομίζω πως οι τροπολογίες οι περισσότερες αφορούν την διαφάνεια, βελτίωση της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε το σύστημα να λειτουργήσει πολύ πιο αποτελεσματικά. Εδώ συμμερίζομαι την γνώμη της Άρων, πιστεύω ότι για να τα καταφέρουμε αυτά θα πρέπει να είμαστε πολύ ρεαλιστικοί. Άρα θα πρέπει να πούμε ότι εφόσον έχει καθυστερήσει τόσο πολύ και ενώ πάμε ένα βήμα μπροστά και ένα βήμα πίσω και μέχρι ότου δηλαδή να κλείσω αυτό το ντοσιέ έχει πάει πίσω τέσσερις φορές γιατί πολλές από αυτές τις τροπολογίες ε, που έχουν υποβάλει τα μέλη και οι ομάδες θα γίνουν πιο εύκολες. Ελπίζω πως θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να διατηρήσουμε το θέμα των τροπολογιών που αφορά την σχετική νομοθεσία γιατί πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι να προβούμε σε μια ενιαία αγορά για την πειθαρχία διακανονισμού δεν ξέρω τώρα ποιο όνομα θα βρούμε, πάντως θα πρέπει να έχουμε αυτή τη φιλοδοξία στην πρότασή μας. Δεδομένου ότι είναι πολύ τεχνικό θέμα, υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς σε συμφωνία σε όλες τις πολιτικές ομάδες και θα μπορέσουμε, ελπίζω, αυτό να τα συζητήσουμε. Οποιοδήποτε από τους μη σκιώδες που ενδιαφέρονται για αυτά τα θέματα, αν θέλει να έχει κάποιο έγγραφο και νομίζει πως δεν το έχει πάρει, παρακαλώ να έρθει σε επαφή με το γραφείο μου ώστε να του δώσουμε αντίγραφα των κειμένων. Δεν είναι τίποτα μυστικό. Είναι όλα κείμενα δημόσια και φαντάζομαι και πως και οι σκιώδεις ε, θα, πιστεύουν το ίδιο, ότι πρέπει δηλαδή να το φτιάξουμε σωστά. Έχουμε έγγραφα τα οποία πρέπει να εξετάσουμε, τα συζητήσαμε και πιστεύω πως μέχρι το καινούριο χρόνο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα. Για τις τραπεζικές υπηρεσίες και πώς θέλουμε να προχωρήσουμε. Ε, πιστεύω πως θα συμφωνήσουμε στις πολιτικές ομάδες. Εγώ θα ήθελα να τα καταφέρω ε, να μην έχουμε διχασμένη πλειοψηφία. Αν μπορούμε να έχουμε πιο ανταγωνιστική διαδικασία διακανονισμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω πως θα είναι πολύ θετική εξέλιξη. Ευχαριστώ πολύ και στόχος είναι να ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 21 Ιανουαρίου του επόμενου έτος και αυτό και να το ψηφίσουμε μετά στην, στην Ολομέλεια του Μαΐου. Οπότε θα έχουμε χρόνο για να κάνουμε τριμερείς διαλόγους και τα λοιπά. Ελπίζω πως θα μπορέσουμε να τηρήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα, γιατί η Κομισιόν είπε να περιμένουμε πως να έχουμε, μέχρι να έχουμε την νομοθεσία περί αξιογράφων. Υπό το φως της εμπειρίας ε, δεν θα ήταν ασφαλές να το αφαιρέσουμε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και προχωράμε στις ψηφοφόρειες που προβλέπονται στις 10.30. Οπότε έχουμε ένα μικρό διαλυματάκι μέχρι τις 10.30. Σας ευχαριστώ. Γεια Καλά λοιπόν, ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας, λέει η Πρόεδρος, και πρώτα θα σας ζητήσω συγγνώμη γιατί πρέπει να προχωρήσω πρώτα στις ανακοινώσεις της Προέδρου, αφού τις ανέβαλα χθες πριν αρχίσει η συζήτηση με τον ε, κύριο Ντράγκη. Τώρα για τις ε, καταξουσιοδότηση, παρακαλώ ησυχία, καταξουσιοδότηση πράξης, παρακαλώ λίγη ησυχία. We won't start the votes until we've got quiet. Um, no, no, no, it's, it's also those two there. Yeah. Okay. Right, first of all, the, the committee... Πρώτα λοιπόν, η Κομισιόν προτίθεται σύντομα να εγκρίνει ε, προτάσεις κατά εξουσιοδότηση στα πλαίσια του ΕΜΙΡ και, τα σχετικά, και τις σχετικές προδιαγραφές που έχουν ήδη υποβληθεί τέλη Σεπτεμβρίου και γι' αυτό η προθεσμία είναι τέλη τούτου του μηνός. Στις 19 Δεκεμβρίου προτίθεται να τα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς τροποποίησης στα σχέδια. Ένα μήνα έχει το Κοινοβούλιο μετά για, τον για την εξέταση των εγγράφων αυτών και γι' αυτό πρέπει... Ωστόσο, είναι πολύ σύντομο στην περίοδο αυτή. Γι' αυτό, εξ ονόματο τη Επιτροπή Οικονομικών, θα ζητήσω παράταση κατά ένα μήνα για την ε, περίοδο ε, κοινοβουλευτικού ελέγχου. Επίσης, η Κομισιόν δεν έχει απαντήσει σε σχόλια που υπέβαλαν μέλη της ΕΚΟΝ για το σχέδιο για τις τεχνικές προδιαγραφές που υποβλήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου, ούτε επίσης σε σχετική επιστολή του εισηγητού Βέρνερ Λάγκεν στα μέσα Νοεμβρίου. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει το δυνατόν συντομότερο, ώστε οι απαντήσεις της να ληφθούν υπόψη στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εν των επεισοδίων αυτών, και επειδή η περίοδος κοινοβουλευτικού ελέγχου πέφτει στα, ε, στην εποχή των ε, διακοπών θα πρέπει να είμαστε και να επαγρυπνούμε περισσότερο σχετικά με τις ε, προθεσμίες για να μην τα επιβάλλουμε αυτά στους ίδιους τους εαυτούς μας διότι γίνεται μέσα σε μια ετήσια βάση και μπορεί τέτοια πράγματα όπως οι πράξεις κατεξουσιοδότηση να είναι όλο και συχνότερες σε όπω όπως MIFID κλπ. Τώρα, για τον τριμερή διάλογο, για τη διαδικασίες τριμερούς διαλόγου, για, το, για την οδηγία και κανονισμό, για τις απαιτήσει κεφαλαίου. Κάναμε δύο διαλόγου, διαλόγους, τρίτη, τρίτη και πέμπτη στο Στρασβούργο και εκεί καλύψαμε ορισμένα σημαντικά θέματα για ε, έξτρα κεφαλαιακά πλαίσια, για την ε, αποζημίωση, η ρευστότητα, και ε, ποσοστό μόχλευσης. Υπάρχουν ορισμένα θέματα ακόμα στην ημερήσια διάταξη, παρόλο που υπάρχουν προσωρινές θέσεις οι οποίες ε, μπαίνουν σε διαπραγμάτευση, σε διμερείς ε, διαπραγματεύσεις την Τετάρτη. Δυστυχώς έγγραφα δεν υπήρχαν για να διανεμηθούν, ούτε εγώ ίδια δεν τα έχω και ελπίζω ότι ένα ενοποιημένο κείμενο των θέσεων μέχρι τώρα θα μπορέσει να συνταχθεί και να διανεμηθεί, έτσι ώστε οι πολιτικές ομάδες αλλά και τα μέλη να είναι ενήμερα. Πρέπει τώρα να θέσω υπόψη σας δύο πράγματα. Πρώτον, Venture Capital Funds και, η Ταμείο Ευρωπαϊκού Επιχειρήν. Είχαμε προχωρήσει συμφωνία με υποδανική προεδρία, όμως εκεί δεν προχώρησε λόγω των φορολογικών και όπως είπαμε στην τελευταία συνεδρίαση έχει επιτευχθεί η πολιτική συμφωνία για τα δύο αυτά θέματα στις αρχές του Δεκεμβρίου και τώρα ε, Σεπτεμβρίου μάλλον και έχουμε επιστολή της 12 η Σεπτεμβρίου γι' αυτό θέτω πάλι υπόψη το θέμα της ε, υπόψη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 73 του κανονισμού και θα δώσω το λόγο σε έναν ή και περισσότερους εκ των εισηγητών. Θέλει να πει κάτι. Φίλιπ Λαμπέρ ή να προχωρήσουμε, εκτός αν κάποιος ενίσταται. Αλλιώς θα κάνουμε την ψηφοφορία στην Ολομέλεια επί του συμφωνημένου κειμένου είτε το Φεβρουάριο είτε το Μάρτιο, αφού το εξετάσουν πρώτα οι νομική νομικοί του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εκτός αν υπάρχουν ενστάσεις. Δεν υπάρχουν, οπότε θα προχωρήσει το θέμα αυτό. Right. Um, το ίδιο πρέπει να γίνει για τους οργανισμούς πιστοληπτικής ικανότητας. Έγινε μια καταρχήν απόφαση τον Νοέμβριο και θέλετε να λάβετε το λόγο. Όχι, μόνο θέλω να επιβεβαιώσω την συμφωνία. Ήτανε, ε, έγινε με κόπο η συμφωνία αυτή οι αφετηρίες του Κοινοβουλίου ήταν διαφορετικές από του Συμβουλίου. Ευχαριστώ ιδιαίτερα πάντως τους σκιώδης ηγητές για τις παρεμβάσεις τους που ήταν ε, κέρυες για τις ε, διαπραγματεύσεις και θα πρέπει να συζητήσουμε στο Στρασβούργο. Νομίζω ότι είναι στις 15 Ιανουαρίου, Τρίτη. Δεν έχω τίποτε άλλο να προσθέσω. Ορισμένα πράγματα τα είπα χθες. Συζήτησα και με τον Κύπριο Υπουργό Οικονομικών. Δεν έχω τίποτε άλλο να προσθέσω. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Εάν δεν υπάρχει ένσταση εκ μέρου μελών της Επιτροπής Οικονομικών, τότε θα επανέλθουν τα κείμενα αυτά τον Ιανουάριο του 2013. Δεν βλέπω ένσταση καμία. Και τέλος, Εθνική και Περιφερειακή Λογαριασμοί, 7 Δεκεμβρίου, συμφωνία με το Συμβούλιο για όλα τα εκκρεμή θέματα σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών και κάτι το οποίο επιτρέπει την εφαρμογή του six-pack. Η τελευταία διαπραγμάτευση έγινε με γραπτή διαδικασία. Οι πολιτικές ομάδες έχουν λάβει τα σχετικά έγγραφα. Εγώ είμαι η συγγήτρια της Επιτροπής μας, επειδή κανείς άλλος δεν προσεφέρθη. Γι' αυτό επαναφέρω το θέμα αυτό υπόψη σας. Στη διάρκεια της εργασίας αυτής διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ακόμη πράγματα τα οποία πρέπει να πιέσουμε να προχωρήσουν και θα το πράξω αυτό είτε με έκθεση ιδίας πρωτοβουλία είτε με ψήφισμα, αλλά αυτά θα συζητηθούν στο πλαίσιο των συντονιστών σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα δηλαδή, διότι οι στατιστικές προφανώς είναι πολύ σημαντικές. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους, ε, νομομαθείς, νομι, τους, ε, τους γλωσσομαθείς νομικούς του ε, Κοινοβουλίου γιατί σε για την εμπειρογνωμοσύνη και πραγματογνωμοσύνες τους, διότι πρόκειται για χιλιάδες ε, σελίδων και θα κληθούν να τα ξανακάνουν όλα αυτά μαζί με το Συμβούλιο πριν να καταλήξουμε στην ψηφοφορία. Άρα δεν έχουμε ακόμη καταλήξει στο πότε θα εγγραφεί στο χρονοδιάγραμμα. Έχετε ένσταση να προχωρήσει σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Δεν βλέπω κανείς να ενίσταται. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για τη συνεργασία σας θα γίνουν ακόμα πιο περίπλοκα με το νέο άρθρο 70 όπως θα δείτε σε λίγο και μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στην έκθεση Φιλίπ Μπάκερ για την βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Α, με συγχωρείτε, μήπως, μήπως προχώρησα πολύ γρήγορα. Όχι, δεν είναι λοιπόν αυτό, είναι πρώτα οι ευρωπαϊκές στατιστικές. συκλούν Είστε έτοιμες και έτοιμοι. Ας κάνουμε πρώτα μια ε, δοκιμαστική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία, πατήστε κάποιο από τα κουμπιά. Ποιο ψηφίζει υπέρ των διακοπών. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ τα κλείνει η ψηφοφορία και έχουμε 34 που θέλουν να πάνε διακοπέ και δύο απόχέ. Τροπολογία λοιπόν 41. Ψήφι υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. Συμβιβαστική α υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. Συμβιβαστική β υπέρ αν με συγχωρείτε, είναι σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος, πρώτο μέρος της συμβαστικής Β υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται αυτό. Προχωρούμε στην τροπολογία 48 υπέρ, κατά, υπέρ, ε, απορρίπτεται. Συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. Αν επιθυμείτε μπορούμε να επαληθεύσουμε. Τροπολογία 55. Απερίφθη, απερίφθη. 17 υπέρ 20 Συμβαστική ε σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική F, σχηματάφτα δηλαδή. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 62 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά είναι καλύτερα να επαληθεύσουμε. Τροπολογία 62. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται λοιπόν με 20 ψήφους υπέρ και 16 κατά. Συμβαστική H σε τρία τμήματα. Πρώτο υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Α, υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Μια στιγμή. Μετά από αυτό. Έντουαρτ, εσεί θέλετε να λάβετε το λόγο. Η προφορική τροπολογία αναφέρεται στο δεύτερο τμήμα που προτιθέμεθα να αλλάξουμε με στενή παρακολούθηση από τα εθνικά κοινοβούλια. Με στενή παρακολούθηση, close monitoring από τα εθνικά κοινοβούλια. Η Ρόδη Κράτσα. Άρα δεν υπάρχει ένσταση για την προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε με την προφορική τροπολογία το ε, τμήμα δεύτερο. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Διακόπτη πρόεδρος. Τροπολογία 71 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά καλύτερα να επαληθεύσουμε. Τροπολογία 71. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. 22 υπέρ 15 κατά. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση, καλώς. 74. Τέλος, 21 υπέρ 17 κατά. Συμβαστική Α Ι, υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 78 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται α, επαλήθευση, καλώς Α, για κοιτάξτε, εγκρίθηκε. 20 υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται επομένω. Συμβαστική J. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18. Υπέρ, κατά, αποχές,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 ξαναβάζουμε τη λέξη harmonized, δηλαδή της λέξης unified. Με την λέξη unified, ψήφι υπέρ, κατά. Ακούω διαφόρους να λένε ναι ή όχι, αλλά δεν υπάρχει ένσταση για την προφορική τροπολογία που επαναφέρει το unified αντί δηλαδή το harmonized. Αν θέλετε το αντίθετο, harmonized αντί unified. Δεν την έχω αυτή την προφορική τροπολογία. Δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς τι σημαίνει λέει η πρόεδρο. Λοιπόν, υπάρχει στο κείμενό σας η λέξη unified, ενοποιημένη. Και τώρα αλλάζει και γίνεται harmonized, εναρμονισμένη. Εσύ λοιπόν καλώς. Ωραία, με το harmonized ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 εκπίπτει. 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, αυτή απορρίπτεται. Προχωρούμε τώρα στην ψηφοφορία του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Αρχι, αρχίστε την ψηφοφορία, ανοίξτε την ψηφοφορία σας παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι, τέλος. 38 υπέρ, μία αποχή και καμία κατά. Τώρα, επί του νομοθετικού περιεχομένου ψηφίσματος, ψηφίσατε όλοι, πέρας 38 υπέρ μια κατά μία αποχή. Η Σοφή, πριν προχωρήσουμε στην τελευταία ψηφοφορία, για την απόφαση να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις συμφωνίας στην πρώτη ανάγνωση, δηλαδή για τη χορήγηση εντολής, θα ήθελα να πω ότι υποστηρίζω απολύτως τον εισηγητή στη διαπραγματεύση Ωστόσο, σημειώνω ότι έκανα και στην προηγούμενη συζήτηση ότι αυτό που εγκρίναμε εδώ, κατά τη γνώμη μου, δεν αποτελεί μια συνεκτική ρύθμιση που να συμβιβάζει την λογοδοσία με τον δημοκρατικό έλεγχο. Είναι μια, ένα μείγμα που περιλαμβάνει λίγο κυβερνήσεις, ε, επικεφαλής στατιστικών ε, υπηρεσιών, ακόμα και το ελεγκτικό συνέδριο και όλοι αυτοί παίζουν διαφορετικούς ρόλους και για μένα ακόμα εξακολουθεί να είναι ασαφές πώς όλοι αυτοί ε, συνεργάζονται. Γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω τον εισηγητή να εξασφαλίσει ότι η έκβαση των διαπραγματεύσεων θα είναι πιο συνεκτική και σαφέστερη, που νομίζω ότι αυτό βρίσκεται στο, είναι προς το συμφέρον της δημοκρατίας. Ποιος εποπτεύει ποιον και ποιος είναι ανεξάρτητος. Ευχαριστώ, Φίλιπ. Συμφωνώ εν μέρη με την Σοφή. Αλλά άλλα τα σπαγκέτι που είπε η ίδια, άλλα τα κανελόνι που είναι απλά. Ή, άμα είναι σκέτα, τους βάζει μια ωραία σάλτσα, γιατί η με σάλτσα μπορεί να είναι και θαυμάσια. Ευχαριστώ. Το πρώτο κείμενο εκών που εγκρίνουμε με τον νέο, με υπό την ισχύ του νέου άρθρου 70 για διαπραγματεύσει σε τριμερή διάλογο. Γι' αυτό πρέπει να ληφθεί τώρα ρητή απόφαση για να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσει που σημαίνουν μια ψηφοφορία. Ψηφοφορία δηλαδή της πλειοψηφίας των μελών της ΕΚΟΝ, όχι των παρόντων μελών. Άρα πρέπει να έχω τουλάχιστον 25 συν, 25 ψήφους υπέρ. Η απόφαση περιλαμβάνει την εντολή, ο συνήθως, για την έκθεση και τη διαπραγματευτική ομάδα που αποτελείται από πρόεδρο, εισηγητή και shadows ή εκπροσώπους, ή εκπρόσωπο μάλλον της πρόεδρου που μπορεί να είναι αντιπρόεδρος, μπορεί να είναι και ο εισηγητής. Ίσως είναι απλούστερο να κάνουμε την ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Η απόφαση λοιπόν για τις διαπραγματεύσεις για συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση και για τη διαπραγματευτική ομάδα. Μένει ακόμα ορισμένοι να ψηφίσουν. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Κλείνω την ψηφοφορία. 38 υπέρ, μία κατά και ουδεμία αποχή. Άρα θα προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις για συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση και θα επανέλθουμε να σας ενημερώσουμε ως συνήθως. Ευχαριστώ πολύ και τώρα προχωρούμε στην έκθεση Φιλίπ Ντεμπάκερ για την βελτίωση της, χρηματο... της ε, χρηματοδότησης των μικρών και μεσών επιχειρήσεων. Ακόμα και ε, δεν είναι απόλυτα η Γραμματεία ξεκινάμε. Αρχικό κείμενο, τίτλος «Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται». 22 ε, «Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται». Συμβιβαστική Α. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική β Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 34 καλύπτεται, 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική C με προφορική τροπολογία που έχει ζητήσει το ΕΛΚ και λέει τονίζει τη σημασία ενίσχυσης του τοπικού τραπεζικού συστήματος. Ε, αντιρρήσεις όχι. Ωραία λοιπόν, τότε ψηφίζουμε με αυτή την προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα το ελέγξω. Είδα κάποια χέρια, αλλά θα το ελέγξουμε. 48. Ε, έλεγχο. έλεγχος. Α, τώρα αλλάξαν κατεύθυνση τα χέρια. Καλό είναι να ελέγχει κανείς. Καλό είναι να ελέγχει κανείς. Λοιπόν, είμαστε πιο σίγουροι. Αρχικό κείμενο. Τίτλος 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. <clears throat> Συμβιβαστική β μάλλον ε, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική F, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται. Συμβαστική FF Υπέρκατα κατά αποχές εγκρίνεται. Τίτλος 3 αρχικό κείμενο, πρωτότυπο κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρκατα κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πρωτότυπο κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 71 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρωτότυπο κείμενο, τίτλος 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 79, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΑΕ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. N υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, παράγραφος 20, υπέρ, μισό λεπτό. Γιατί λέει να πας στα 107. Α, ναι, σωστά, το κάναμε αυτό. Παράγραφος 20. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τίτλος 6. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 109. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 111. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πρωτότυπο κείμενο της παραγράφου 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 112 έχει αποσυρθεί. 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Θα το ελέγξω ηλεκτρονικά γιατί κάτι παράξενο μου φαίνεται. It's closed and it was carried 23 16. Um, Εγκρίθηκε 23 προς 16. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχέσεις απορρίπτεται. 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πρώτο, παράγραφος 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική ο μικρόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 127 υπέρ κατά αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 127. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. 128 έχει καλυφθεί, 129 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 131 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 132 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Να το ελέγξω το 132. Νομίζω πως το ΕΛΚ ήταν μόνο του. Τέλος ψηφοφορίας. Να, 22 υπέρ, 17 κατά. 135 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 136 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 140 υπέρ που είναι ένα εκτιμώντας υπέρ κατά να ελέγξουμε την 140 Τέλος πληροφορία και καταπίπτει. Εκτιμώντας ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εν, τροπολογία ένα υπέρ αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία δύο. Μπορούμε να τα κάνουμε unblock εκτός από τη 4. Ωραία λοιπόν. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Έχουμε κάνει λοιπόν όλα τα εκτιμώντας και πάμε στη συμβιβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εκτιμώντας α τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εκτιμώντας C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 18 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα πάμε στην τροπολογία της Επιτροπής Απασχόλησης. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε για αυτήν παρακαλώ 24 της Επιτροπής Απασχόλησης. 41 είναι οι μάλιστα. Απορρίπτεται 19 υπέρ 22 κατά. Ήμκο 14 υπέρ. Κατά αποχές. Ας ελέγξουμε τη 14 της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς. Ψηφίζουμε ΙΜΚΟ 14. Ψηφίσατε όλοι αυτό που θέλατε. Ωραία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 21 προς 19. Ήμκο 23 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Ήμκο 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τέρμα. Ψηφίζουμε τώρα για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά. Voted. Ψηφίσατε όλοι. Κλείνει η ψηφοφορία. 39 υπέρ, μια κατά, καμιά αποχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν φτάσαμε στις ευχές ακόμη. Oh, I see. Right. So that's 40 in favor. Okay, right. Εντάξει, τότε είναι 40 υπέρ. Δεν δούλεψε η κάρτα, μάλλον. Meeting is the 10th of January. 10 Ιανουαρίου είναι η επόμενη μας συνεδρίαση. Καλές σας διακοπές και καλά Χριστούγεννα. Φιλίπε, έχουμε ήδη εικόνα για το χρονοδιάγραμμα των διαφόρων τριών μερών διαλόγων στην εβδομάδα 7 Ιανουαρίου. Δεν μπορώ να στο πω αυτό χωρίς να δω και που λέει για τον τριμερή διάλογο.